να καλωσορίσω την κυρία Βιολέτα Μπούλτς, την Επίτροπο λοιπόν, που θα μας κάνει την ανακοίνωση για την μελλοντική δέσμη για τις αερομεταφορές. Η κυρία Μπούλτς έχει το λόγο. Θα δώσουμε επίσης το λόγο ε, ή μάλλον θα δώσουμε αμέσως το λόγο στην Επίτροπο και μετά από την παρουσίαση της Επιτρόπου θα ακολουθήσει η συζήτηση. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι ενώπιόν σας σήμερα για να συζητήσουμε τη μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές. Μου αρέσει πολύ το ενδιαφέρον που δείχνετε για το θέμα και χαίρομαι που βλέπω ότι οι εκτιμήσεις μας επικαλύπτονται σε πολλές ε, περιπτώσεις. Όσοι γνωρίζετε, οι αεροπορικές μεταφορές είναι σημαντικός μοχλός για την ανάπτυξη οικονομίας, για την ανταγωνιστικότητα και το καθεξής. Για την απασχόληση, γι' αυτό η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στον τομέα αυτό παίζει κέριο ρόλο για την ευρωπαϊκή οικονομία και για τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την ηγετική της θέση προς το συμφέρον των πολιτών της και των ε, επιχειρησιών της. Ικανοποιεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η στήριξη που δίνεται στην έκθεσή σας και η σημασία που αποδίδεται στην αεροναυτική βιομηχανία για την καινοτομία, για την προσφορά υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Για έναν δηλαδή ανταγωνιστικό και βιώσιμο τομέα αεροπορικών μεταφορών. Συμφωνούμε μαζί σα που ζητείτε να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον τομέα αεροπορικών μεταφορών. Η επικείμενη στρατηγική, δηλαδή αυτή που πρόκειται να κατατεθεί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη στι 2 Δεκεμβρίου, θα αποτελέσει την συμβολή μα στην προσπάθεια διαμόρφωση του μέλλοντος των αεροπορικών μεταφορών μέσα σε ένα συνολικό σε μια συνολική προσέγγιση ή αν θέλετε μια ολιστική προσέγγιση. Ό,τι αφορά τι συγκεκριμένες ε, τα συγκεκριμένα αιτήματα και μια και συνεχίζεται στην πραγματικότητα η δουλειά μα, επιτρέψτε μου να τονίσω πρώτα ορισμένα θέματα. Πρώτα, μια παγκόσμια προοπτική. Η παγκόσμια αγορά αεροπορικών μεταφορών βρίσκεται σε φάση αλλαγών. Να μην φοβούμαστε όμως τις αλλαγές αυτές. Να τις συνοδεύσουμε, να παίξουμε μίζωνα ρόλο στην διαμόρφωση αυτού του νέου κόσμου στις αεροπορικές μεταφορές. Στα πλαίσια αυτά, συμφωνώ μαζί σας, ότι είναι κρίσιμο για την αεροπορική βιομηχανία να είναι καλά εξοπλισμένη για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους άλλους σημαντικούς φορείς όπως για παράδειγμα από την Ασία και την Μέση Ανατολή. Μόλις επέστρεψα σήμερα από την Μέση Ανατολή και σας βεβαιώνω ότι είναι απόλυτα αληθές αυτό που ισχυρίζομαι. Με την επιδίωξη φιλόδοξης εξωτερικής πολιτικής αεροπορικών μεταφορών μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύναψη ε, συμφωνιών ε, με σημαντικές αγορές για την πρόσβαση στις αγορές αυτές για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προωθήσει τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αξίες της και θα αποτρέψει τις στρεβλώση του ανταγωνισμού. Χαίρομαι που ζητείτε και εσείς τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ε, πρακτικών αθέμητου ανταγωνισμού στην διεθνή αεροπορική ε, συγκοινωνία. Γι' αυτό και λαμβάνει νέα μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αθέμητες ανταγωνιστικές πρακτικές από τρίτες χώρες και από τους operator, ε, operator επιχειρηματίες δηλαδή των τρίτων χώρων. Επίσης, δεύτερο τώρα, η ενιαία αγορά. Από τη σκοπιά της ενιαίας αγοράς βλέπουμε ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείε εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, άλλες όμως τα πάνε πολύ καλά. Εξάλλου, Ορισμένα μεγάλα αεροδρόμια αποκομίζουν σημαντικά κέρδη από τι του, αλλά μικρά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν προβλήματα. Συνολικά τα πάμε καλά. Ωστόσο, δυστυχώ η εικόνα είναι μάλλον μεικτή. Εν ώψη αυτού του ιστορικού, εμεί εξετάσαμε προσεκτικά το ρυθμιστικό πλαίσιο τη Ένωση. Γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαίε και άλλε βελτιώσει έτσι ώστε το τομέα να γίνει πιο αποδοτικό να προσφέρει σταθερότητα στους επενδυτές, να ενθαρρύνει την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη και βεβαίως να διατηρήσει σε πολύ ψηλό επίπεδο την ασφάλεια. Τρίτο, η Άσα. Είμαι πεπισμένη ότι οι προτάσεις για τον, την αναθεώρηση του βασικού κανονισμού της ΕΑΣΑ θα της επιτρέψει να συνεχίσει να παίζει το ρόλο της και με τη συμμετοχή βεβαίως των πολιτών του κλάδου και των ε, νομοθετών, των ρυθμιστών δηλαδή, να εισαχθούν νέοι μηχανισμοί για, για εποπτεία ασφάλειας και για κανόνες που είναι βασισμένοι στην αποδοτικότητα. Στην αναθεώρηση θα καταστρώσουμε το πλαίσιο και για την λειτουργία, τη ρυθμίση της λειτουργίας δηλαδή όλων των μη επανδρομένων αεροσκοφών στην Ευρώπη. Συγχαίρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έργο του στην έκθεση για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Κοινωνικά θέματα. Πολλά τέτοια κοινωνικά θέματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στις αεροπορικές συγκοινωνίες και να διατηρήσουμε ένα εργατικό δυναμικό με υψηλά προσόντα και δεξιότητες. Ταυτόχρονα τα επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν προκύψει και έχουν επιπτώσεις στην απασχόληση πρέπει και αυτά να εξεταστούν προσεκτικά. Ένας σε βαθο κοινωνικός διάλογος είναι απολύτως αναγκαίος. Πέμπτο, βελτιώσεις και καινοτομία. Τονίζετε εσεί την σημασία της εφαρμογής του Ενίου ευρωπαϊκού ουρανού που θα επιτρέψει τον εξυγχρονισμό της διαχείρισης των ε, ροών των αεροπορικών συγκοινωνιών και καλύτερη βέβαια επιτήρηση των υπηρεσιών και επιτρέπει την βελτίωση της ικανότητας λιγότερες εχμές και καθυστερήσεις και μείωση του κόστους για τον τομέα των αεροπορικών συγκοινωνιών. Σε ό,τι αφορά το ΣΕΖΑΡ, έχουμε τώρα ένα πλέον συνεκτικό project με ξεκάθαρο πλαίσιο, με καινοτόμες εταιρικές σχέσεις με κίνητρα που είναι σε θέση να προωθήσουν νέα κόνσεπτ για την διαχείριση. Συμφωνούμε λοιπόν με την επιθυμία σας να εφαρμοστούν όλα αυτά το δυνατόν συντομότερο. Για το λόγο αυτό απηχώ και την δυσαρέσκειά σας για τα ελλείμματα στην νομοθεσία, τα σλότ, ο ενιαίος ε, ε, ευρωπαϊκός ουρανός, τα δικαιώματα των επιβατών. Η πολιτική σας στήριξη εκτιμάται πάρα πολύ από εμάς. Έκτο, το περιβάλλον. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις επιπτώσεις των περιβάλλον ενός τομέα που βρίσκεται σε ανάπτυξη. Χρειάζονται λοιπόν καινοτόμες σύγχρονες λύσεις για να μειωθεί το αποτύπωμα στο δικτύο του άνθρακος του τομέα. Τα είπα στα, στις αεροπορικές εκθέσεις του Παρισιού και του Ντουμπάι. Η τεχνολογία είναι υπηρέτης μας. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ισχυρά ρυθμιστικά εργαλεία για να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Ο ΔΕ θα πρέπει να παίξει ένα κρίσιμο ρόλο στην ε, εξέβρεση μιας παγκόσμιας λύσης. Εμείς θα κάνουμε κάθε τι που περνά από το χέρι μας για να τον διευκολύνουμε. Πιστεύω ότι ε, με συνεργασία μαζί σας μπορούμε να εξασφαλίσουμε έναν ισχυρό κλάδο ευρωπαϊκών αεροπορικών συγκοινωνιών και αναμένω με ενδιαφέρον τις απόψεις σας. Ευχαριστώ την κυρία Βιολέτα Μπούλτς, την Επίτροπο Βιολέτα Μπούλτς. Θα ξεκινήσουμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Μαρινέσκου δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, όπως είπε και η Επίτροπος ήδη, αυτός ο τρόπος, ε, ε, αυτός ο τομέας μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικός για την οικονομία, για την απασχόληση. Δεν μπορούμε ε, να διανοηθούμε το μέλλον μας χωρίς τις αερομεταφορές βλέπουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα όταν ε, γίνεται απεργία σε αυτό το κλάδο και γι' αυτό θα πρέπει να τον υποστηρίξουμε από όλες τις πλευρές ε, υποδομές ε, των αερολιμένων, ε, περιφερειακά αεροδρόμια, νέες υποδομές διότι τις χρειαζόμαστε εξασφάλιση των αεροπορικών εταιριών, δηλαδή να ισχύουν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού, βάσει των οποίων θα λειτουργήσουν και σε συνεργασία με άλλες περιοχές του κόσμου για να επικρατήσουν εναρμονισμένα πρότυπα. Ελπίζω να ε, έχετε σύντομα και τη διαπραγματευτική εντολή για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ε, με τις ε, χώρες του κόλπου. Για το SES 2 e το χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε το CISAR, την εφαρμογή του σε μία νέα όμως αρχιτεκτονική, όχι στην τρέχουσα. Αλλιώς θα χάσουμε πολλά κονδύλια και πάρα πολύ χρόνο. Σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να σεβαστούμε τον διεθνή οργανισμό και το ρόλο που τη αναλογεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος και στο Συμβούλιο, όπου υπάρχουν προς το παρόν κολλήματα, και να ε, επαναλάβουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριο Ερτούκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Θίξατε πολλά, κυρία Μπούλτς, από αυτά που έχουμε συζητήσει και εμάς. 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι στον κλάδο αεροπορικών ε, συγκοινωνιών. Και τζίρο 360 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Μεγάλη σημασία του κλάδου αυτού. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τη διεθνή μας ανταγωνιστικότητα. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Σήμερα συζητούμε πράγματα τα οποία ζητούμε να δούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Aviation Package. Γνωρίζουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικό ανταγωνισμό διεθνώς. Ανταγωνισμό που χαίρει και κρατικών ενισχύσεων. Είτε πρόκειται για τις χώρες του Περσικού κόλπου, είτε για χώρες της Ασίας. Παρ' όλα αυτά, ως απάντηση να μην αντιδράσουμε με προστατευτισμό, να επιλέξουμε καλύτερα μια ευφυή στρατηγική, να επιζητήσουμε την συνεργασία στη βάση της διαφάνειας και της εντιμότητας. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την αναθεώρηση της οδηγίας 868 του 2004 και εσωτερικά να κάνουμε το καθήκον μας, έτσι ώστε, δηλαδή εντός της Ένωσης, ώστε να μπορούμε να επιδιώξουμε στόχους και προς τα έξω. Θα ήθελα να έρθω τώρα στις κοινωνικές πτυχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίσατε και εσείς κυρία Επίτροπε ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους καλά εκπαιδευμένους και να έχουν διάθεση να εργαστούν. Αυτά βεβαίως χρειάζονται βελτίωση οι συνθήκε εργασία του χρειάζονται βελτίωση. Άρα, να κάνουμε πρώτα το καθήκον μας εδώ, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά να προχωρήσουμε σε διεθνεί συμφωνίε. Ευχαριστώ. Φώστερ, παρακαλώ. Δυο λεπτά. Στο όνομα βέβαια της ομάδας ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει και θα επικεντρωθώ στο περιεχόμενο. Ε, της έκθεσης. Ε, φυσικά ε, έχουμε σε ένα ορισμένο βαθμό διακομματική συμφωνία. Όσο επιτοπλίστων συμφωνούμε με το περιεχόμενο. Δυστυχώ όμω τρία είναι τα σημεία που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Καταρχά ε, η αναφορά στα θέματα ανταγωνισμού. Δεν είναι ο ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου, να αποφασίζει πώς, τι θα κάνουν οι αεροπορικέ εταιρείε στι τρίτε χώρε με τη χρηματοδότησή του. Ε, αυτό είναι θέμα συμβάσεων, θέμα διεθνών υποχρεώσεων. Δεν είμαστε σε θέση εμεί να παρεμβαίνουμε. Ε, αυτή η προσέγγιση σίγουρα θα πλήξει και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής όσο και της δραστηριότητα των αεροπορικών μας εταιριών. Δεύτερον, το κεφάλαιο για το κοινωνικό θεματολόγιο. Τονίζουμε ότι ε, ε, ε, υπάρχει διαρκής ανάπτυξη στον κλάδο και Χρειάζεται υψηλή ειδίκευση και υπάρχουν ε, ισχυρά κίνητρα για τους εργαζόμενους. Ε, υπάρχει προστασία για τα κοινωνικά πρότυπα, για τη συλλογική διαπραγμάτευση και θα πρέπει να διατηρηθεί η προστασία που υπάρχει. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και άλλες παράγραφοι οι οποίες είναι εξαιρετικά ε, περιοριστικές σε σχέση με τον τρόπο προκήρυξης της θέσης, με τους όρους εργασίας που δεν συμβαδίζουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ΕΤΡΑΝ. Στη συνέχεια μιλάμε για το ρόλο της ΕΑΣΑ στον ε, ΙΚΑΟ και αναφέρουμε ότι είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός διεθνής οργανισμός. Εμείς δεν υποστηρίζουμε μια ευρωπαϊκή φωνή σε αυτό το τομέα, διότι υπάρχουν πολλές χώρες που βάσει τη σύμβαση του Σικάγο ανήκουν άμεσα στον ΙΚΑΟ, οπότε δεν θα θέλαμε να καταργηθεί ο εκπρόσωπος κάθε χώρα ε, στον ΙΚΑΟ. Και τέλος, Πρόεδρε, για αυτούς τους λόγους έχουμε καταθέσει χωριστό ψήφισμα από πλευρά των συντηρητικών και δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το κοινό ψήφισμα. Παρ' όλα αυτά, ε, περιμένουμε με ανυπομονησία τις προτάσεις ε, της Επιτροπής το Δεκέμβρη. Ευχαριστούμε. Μαΐσνερ για τους ε, φιλελεύθερους. Δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης την Επίτροπο για την ε, παρουσίαση του θέματος και βεβαίως για τις εντυπώσεις που μετέφερε από τις χώρες του Περσικού. Διότι βεβαίως ο κλάδος των αεροπορικών συγκοινωνιών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ευρώπης, άλλωστε εξαρτώνται πολυπληθέστατες ε, θέσεις απασχολήσεως από τον, ε, τον κλάδο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να τον διατηρήσουμε σε καλή υγεία. Έχουμε διάφορα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερη καινοτομία. Πρώτον, νέες ενέργειες, για παράδειγμα νέα υλικά, προτριετίας παρακολούθησα μια παρουσίαση για το αεροσκάφος του μέλλοντος που θα έχει νέα συστήματα τα οποία θα διευκολύνουν. Ε, Βεβαίω πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες στην έρευνα. Χρειαζόμαστε επίσης αεροσκάφη που να είναι πολύ λιγότερο θορυβόδη. Χρειάζεται επίσης να γίνει προσπάθεια να ε, μπορούν οι άνθρωποι που πετούν πολύ να κινούνται ευκολότερα από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο και χωρίς ε, τόσους πολλούς ελέγχους. Βεβαίω, και οι χώρε του Περσικού κόλπου αλλά και ε, άλλοι ανταγωνιστέ δυσχεραίνουν το έργο των αεροπορικών εταιριών της Ευρώπης. Μας είπαν ήδη ότι πρέπει να επαναξετάσουμε τον κανονισμό 868 του 2004 και να δούμε αν είμαστε καλά εξοπλισμένοι κατά του αθέμητου ανταγωνισμού με τον τρόπο αυτό. Ασφαλώς είμαι υπέρ. Ωστόσο θεωρώ ότι πρέπει ακόμη να εξετάσουμε, διότι δεν έχουμε μόνο τις αεροπορικές εταιρείε, έχουμε και θέσεις εργαζομένων στα αεροδρόμια. Επίσης και στην βιομηχανία που παράγει αεροσκάφη. Όταν θα γίνει λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν, χρειάζεται να προσφέρει μια ισορροπημένη θέση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλους τους τομείς αυτούς. Αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει και με συμφωνίες για τις αεροπορικές συγκοινωνίες και αυτό λέχθηκε ήδη. Ορισμένα σχόλια ακόμη. Οι συνθήκες εργασίας ασφαλώς και είναι σημαντικές. Χρειαζόμαστε ελκυστικές θέσεις απασχολήσεως, χρειαζόμαστε διαρκή κατάρτιση, βεβαίως και για τους επιβάτες και για τα πληρώματα χρειαζόμαστε και συνθήκες ασφαλείας. Χρειαζόμαστε ε, δορυφορικά συστήματα που να εντοπίζουν τα αεροσκάφη αμέσως εάν αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα και βεβαίω και τα μικρά αεροσκάφη. Ω απολύτω τελευταίο σχόλιο έχω να τονίσω το εξή. Χρειαζόμαστε βεβαίω ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Το τονίσαμε αυτό και πάνω σε αυτό θα εργαστούμε και ελπίζω να το επιτύχουμε στο μέλλον. Σα ευχαριστώ. Λόπεθ Μπερμέγιο. Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα στο όνομα τη Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς στην θεματολογία ε, της, ε, των αεροπορικών μεταφορών αλλά σε κοινωνικό επίπεδο. Ε, από τη μία έχουμε τους καταναλωτές, από την άλλη έχουμε και τους παραγωγούς, αυτούς που εργάζονται στον τομέα των αερομεταφορών και δυστυχώς εκεί δεν υπάρχουν κέρδη για την ζωή. Είναι ένας από τους τομείς ο οποίος θίγεται περισσότερο από το λεγόμενο κοινωνικό ντάμπινγκ, αυτό επηρεάζει και την ασφάλεια, όπως δείχνουν οι τελευταίες μελέτες και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα πρέπει να αφήσουν να εμβαθυνθεί η φιλελευθεροποίηση του τομέα ε, εις βάρος των εργαζομένων και των επιβατών. Δυστυχώς τέτοια προβλέπουν συμφωνίες όπως το ΤΙΣΑ και άλλα. Θα πρέπει επίσης να μην αμφισβητηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να μην επιβληθεί μείωση των επιπέδων προστασίας των συνθήκων εργασίας. Είδαμε τι συνέβη στη Γαλλία με την ΕΦΑΝΣ. Δεν θέλουμε τέτοιου είδους, θα έλεγα, μέτρα. Θέλουμε να, παραμείνει στο δημόσιο, να παραμείνουν στο δημόσιο οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις και να μην υπάρξει μια πίεση για την ιδιωτικοποίησή τους. Είδαμε τι συμβαίνει επίσης και με περιπτώσεις όπως η ΑΕΝΑ στην Ισπανία. Είναι ένα σκάνδαλο και κοινωνικό και οικονομικό το οποίο επιτελέστη με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και για το περιβάλλον επίσης είναι σαφές ότι οι αερομεταφορές μολύνουν και στη συνάντηση των Παρισίων πρέπει να τεθεί το θέμα. Τρία λεπτά, τέλει, για τους πράσινους. Πραγματικά έχετε πάρα πολύ χρόνο, τρία ολόκληρα λεπτά. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι αερομεταφορές ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ανά αν το πάρουμε και ένα χιλιόμετρο, είναι τρεις φορές πιο επιβλαβή τα αέρια σε σχέση με το αυτοκίνητο από, το Λονδίνο μέχρι τη Νέα Υόρκη, παραδείγματος χάρη. Έχουμε ε, εκπομπές αντίστοιχες με τη θέρμανση ε, ε, ενός έτους για ένα άτομο και πολύ παράξενο δεν υπάρχουν φόροι. Κανένας φόρος για την κυροζήνη και για τις διασυνοριακές πτήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι πρωταθλήτριες για τα φορολογικά δωράκια. Ε, μα είναι όλα ανάποδα. Είναι δυνατόν το μοναδικό ρηκτό κάψιμο που δεν φορολογείται να είναι η κυροζήνη γιατί ε, ε, υπερφορολογείται το πετρέλαιο ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ε, και από το 90 διαρκώς μειώνεται η τιμή των αεροπορικών εισιτήριων ενώ έχουν αυξηθεί κατά 110% οι εκπομπές ε, αερίων και μπορούν μέχρι το 2050 να τριπλασιαστούν, να οι δύο βαθμοί τη υπερθέρμανση. Ε, εκτό αν αλλάξει κάτι στην COP21, ε, Α ε, φορολογήσουμε το καύσιμο επιτέλου, όπω όλα τα υπόλοιπα και να εφαρμόσουμε και για τι αεροπορικέ εταιρείε τον ελάχιστο συντελεστή. Άλλη πρόκληση κοινωνικού χαρακτήρα. Ζούγκλα είναι. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας σε μηδενικές ώρες ψευδής ε, ε, μισθωτή ε, που είναι ανεξάρτητη ε, εικονικές εταιρείες. Ε, επίτροπε που σας έχω εμπιστοσύνη. Μας είπατε τον περισμένο Ιούνιο ότι δεν πρόκειται να ε, εθελοτυφλείτε και ότι θα αρχιεσχολείστε με όλα αυτά τα προβλήματα. Ε, λοιπόν, να ασχοληθείτε με αυτά τα κοινωνικά ζητήματα διότι είναι εις βάρος των εργαζομένων. Πρέπει να αναθεωρήσετε τον 868 του 2014 που ποτέ δεν εφαρμόστηκε

κατά των αθέμητων ως προς ε, την τιμολόγηση. Ryanair, Norwegian Airlines, ε, ε, τέτοιες αεροπορικές εταιρείες πρέπει να υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με το δίκαιο. Αυτός ο κανονισμός πρέπει να μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Εμμυράτων και των αεροπορικών τους εταιριών. Δεκάδες δισεκατομμύρια ενισχύσεις παίρνουν αυτέ οι εταιρείε, Μα πώς εμείς να παρακολουθήσουμε, δεν γίνεται. Χρειάζεται νέος κανονισμός ε, κατά των αθέμητων όρων ανταγωνισμού που στρεβλώνουν την κατάσταση ως προς την τιμολόγηση και τα τέλη. Ε, ε, το κλίμα, τα κοινωνικά ζητήματα και η διεθνής διάσταση. Αυτές είναι τρει τρεις βασικές προκλήσεις. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα. Δεν αναφέρεται τίποτα για αυτά μέσα στο ψήφισμα του ΕΛΚΑ. Εμείς αντίθετα στο δικό μα χωριστό ψήφισμα να δίνουμε απαντήσεις γιατί ο πλανήτης, οι εργαζόμενοι ε, και οι καταναλωτές ε, θα πληρώσουν το μάρμαρο αν δεν κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντέλη. Ε, Αγιούτο, ένα λεπτό έχετε εσείς μόνο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η καλύτερη ευρωπαϊκή επιχείρηση των τελευταίων πέντε χρόνων, σύμφωνα με τη Skytrax, δεν είναι από ένα κράτος μέλος αλλά είναι η Turkish Airlines. Ο κόσμος αλλάζει και ε, όλο και περισσότερο το κέντρο και το βάρος των αερομεταφορών μεταφέρεται προς την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πλέον είναι η Emirates, η Qatar, η Etihad και τώρα πια και η Turkish. Δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας την αποτυχία των ευρωπαϊκών στρατηγικών. Βλέπουμε επίσης ότι στην αεροβιομηχανία μας υπάρχει μια έντονη παρουσία των ξένων κεφαλαίων. Υπενθυμίζω αυτά τα οποία έχει περάσει η εθνική μας επιχείρηση, η οποία θεωρήθηκε σαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την κυβέρνηση Ρέντζη που επειδή πουλήθηκε στην Etihad. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Έχουμε μια εξασθενημένη βιομηχανία καθόλου ανταγωνιστική που δεν διασφαλίζει ούτε τις κανονικές ε, ροές πτήσεων, ούτε τα κέντρα ε, των ε, συγκοινωνιών των αεροπορικών, ούτε τις τοπικές συνδέσεις. Λοιπόν, θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε και να θεωρήσουμε την αρνητική αυτή πορεία σαν αναπόφευκτη. τού. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα καχύποπτη σε σχέση με τους νέους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις έχω την αίσθηση ότι με, με το άλοθη απλοποίησης δημιουργούμε ένα τεράστιο πράγμα το οποίο δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Εμείς ε, οι προτάσεις που κάνει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκουμε ότι έχουν κάποια θετικά σημεία στον τομέα της ασφάλειας. Σαν παράδειγμα έχουμε, είμαστε υπέρ της ενίσχυσης της ασφάλειας. Υπάρχει το θέμα της αεροβιομηχανίας την οποία γνωρίζω καλά ε, γιατί εργάστηκα στην ΕΦΑΝΣ 35 χρόνια και το θέμα της ασφάλειας λοιπόν είναι καθοριστικό Πρέπει να ληφθούν λοιπόν μέτρα εδώ για την ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού των αερομεταφορέων μετά και από το δράμα της German Wings. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και δεν πρέπει να μείνουμε αμέτωχοι βλέποντας στην ουσία να βυθίζονται οι μεγάλες εθνικές αερομεταφορές. Ε, οι μεγάλοι εθνικοί οι προσπάθειες πρέπει να γίνουν από όλους και τους εργαζομένους. Αλλά οι επιχειρήσεις μας δεν θα επιβιώσουν εάν δεν μπορέσουν να ανταγωνιστούν ισότιμα τους ανταγωνιστές τους, δηλαδή τις εταιρείες των χωρών του κόλπου και της Τουρκίας που επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους για να μην μιλήσω για έμεση βοήθεια όπως σχεδόν δωρεά καύσιμα, επιδότηση των κοινωνικών παροχών, ε, όλα αυτά επιβαρύνουν βέβαια τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δεν μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε βοήθεια διότι απαγορεύεται η βοήθεια προς τις επιχειρήσεις στο όνομα ε, του ίδιου του ανταγωνισμού. Συστήνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τη μείωση ε, του ποσού των καυσαερίων, στην ουσία επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις μας και να δημιουργήσετε προβλήματα στους ε, επιβάτες, γιατί θα υπάρξει από τους επιπλέον φόρους αύξηση της τιμής ε, του κομίστρου. Ο κύριος Επιτίδιος, ένα λεπτό παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε στο άμεσο μέλλον να εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα οικονομικής αναπτύξεως των κρατών της ευρωπαϊκής ενώσεως. για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει η σχετική στρατηγική της ευρωπαϊκής ενώσεως να τροποποιηθεί ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. κατά πρώτον ο κλάδος θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστικός για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται από αεροπορικές εταιρείε κρατών που δεν ανήκουν στην ευρωπαϊκή ένωση. σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η αντιμετώπιση του αθέμητου ανταγωνισμού η αναβάθμιση της ασφάλειας των πτήσεων και τέλος ε, η δυνατότητα να υιοθετηθούν τεχνολογίες υψηλής προδιαγραφής και φιλικές προς το περιβάλλον. θα πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και το προσωπικό που εργάζεται στις αεροπορικές εταιρείες να είναι υψηλών προδιαγραφών και να έχει τη δυνατότητα να αφομοιώσει τις ε, σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις τέλος θα πρέπει και τα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα ούτως ώστε να ενισχύσουν τις προσπάθειες που προανέφερα. Ευχαριστώ τον κύριο Επιτίδιο. Ο κύριος Βάντεν Κάμπ έχει το λόγο. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ βεβαίως πρώτα τον κύριο Μαρινέσκου αλλά και άλλους ε, συναδελφούς όπως την κυρία Μάισνερ. Σας ευχαριστώ διότι με τη συνεργασία όλων κατορθώσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συντάξουμε ένα ξεκάθαρο ψήφισμα για τον τομέα των αεροπορικών συγκοινωνιών. Έχω μάλιστα να δηλώσω το εξή, κύριε Πρόεδρε. Οι προσδοκίες τη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο είναι πολύ υψηλές. Θέλουμε πραγματικά στις 2 Δεκεμβρίου να καταλήξουμε σε μια καινοτόμο και φιλόδοξη πρόταση. Θέλουμε να είναι ξεκάθαρη η βάση στην οποία θα μπορέσει να στηριχτεί η κυρία Μπούλτς στις διαβουλεύσεις της με την ε, βιομηχανία, τον κλάδο δηλαδή αεροπορικών συγκοινωνίων στο μέλλον. Ανταγωνιστικότητα. Πρώτα-πρώτα. Η ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία είναι μικρή. Πρέπει ωστόσο να ανδρωθεί και πρέπει να είναι ε, ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Και χρειάζεται έντιμος ανταγωνισμός και από όλους τους ε, εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και ενώ ιδίω εδώ τις χώρες της Ανατολής. Υπάρχουν και εξελίξεις ε, με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη καθώς και με τα δορυφορικά συστήματα. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι το καθημερινό της ψωμί. Ένα τρίτο θέμα, κύριε Πρόεδρε, αναφέρομαι στα όσα είπε ο κύριος Ερτόγκ εδώ, είναι η κοινωνική ατζέντα. Καμιά φορά είναι βαθιές οι τομές που γίνονται ε, στον κλάδο. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, η ασφάλεια. Τα είδαμε με την πτώση του ρωσικού αεροσκάφους, ε, αεροσκάφους στην Αίγυπτο. Η ασφάλεια στην, ε, στις αεροπορικές κοινωνίες είναι μια τεράστια πρόκληση. Η κυρία Αιάλα Σέντερ. Παρακαλώ. Έχει το λόγο. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μέχρι τέλους του έτους θα εγκρίνετε την δέσμη και θα την υποβάλλετε. Πρέπει να σκεφτείτε όλα τα σχετικά με τις αεροπορικές εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Ενέργειο Χώρο. Και να υπερασπίσετε τις ευρωπαϊκές εταιρείε και τους ευρωπαίους επιβάτες απέναντι στις ε, εταιρείε εκείνες οι οποίες δεν τους συμπεριφέρονται καλά. Μην ξεχάσετε και το μεγάλο αριθμό των απασχολουμένων στον κλάδο, καθώς επίσης τους νέους οι οποίοι δεν πληρώνονται καλά. Λοιπόν, να ε, λάβετε υπόψη όλες αυτές τις επιπτώσεις, να λάβετε υπόψη επίσης την ανάγκη να έχουν πρόσβαση στην αγορά και τα μικρά και περιφερειακά αεροδρόμια. Ο κλάδος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ας μην το λησμονούμε. Ευχαριστώ. Πορέμπα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, αντιμετωπίζουν πάρα πολλέ προκλήσει οι αεροπορικέ εταιρείε ω προ την ανταγωνιστικότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτε χώρε. Εμεί προσπαθούμε να επιβάλλουμε ρυθμίσει και περιορισμού, όπω παραδείγματο χάρη το εμπόριο εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκάθαρα αποδυναμώνει τη θέση των αεροπορικών ε, εταιριών. Η πρόταση του Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελπίζω να ε, περιλαμβάνει μέτρα που θα ενισχύσουν ανταγωνιστικότητα και θα έχουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική αναπτυξιακή για τους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των περιφερειακών αεροδρομίων όπως στην περιοχή μου, στη Γιασόνκα παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα μικρό περιφερειακό αεροδρόμιο που είναι δεύτερης ε, κατηγορίας ε, προς το παρόν, όμως θα μπορούσε να αναδειχθεί σε ένα σημαντικό αεροδρόμιο για να αποφορτήσει την κατάσταση στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της ε, Πολωνίας. Περιμένουμε την πρότασή σας ούτως ώστε με στρατηγικό τρόπο να συμβάλετε στην ανάπτυξη του κλάδου και στο μέλλον των αερομεταφορέων. Ευχαριστούμε. Ε, ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό πάλι ο κύριος ε, Τελειώκα. Δυσκολεύονται οι διερμηνείς ε, να σας παρακολουθήσουν τόσο γρήγορα που μιλάτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Μα, μα, είπατε ότι σας ικανοποιεί το ψήφισμα αυτό τι σημαίνει ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση και θεωρούμε ότι είναι εν πάση περιπτώσει ισόρροπη προσέγγιση, δεν είναι τέλεια αλλά αντιμετωπίζει μια, κάποια από τα βασικότερα ζητήματα. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, η δύσκολη κατάσταση των αερομεταφορέων δεν οφείλεται σε λάθη των κρατών μελών. Πάντοτε τα ρίχνουμε όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα χρειαζόμαστε ένα πακέτο για, τους αερομεταφορές Σίγουρα θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς ε, και να ισχύουν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, αλλά η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο προστατευτισμός. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Ε, Επίτροπε και εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία. Αυτά τα 7 σημεία που εκθέσατε κατά τη γνώμη μας ε, θα είναι μια κρατεά βάση για τις ε, μελλοντικέ διαπραγματεύσεις για τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να έχουμε πραγματικό ανταγωνισμό όχι προστατευτισμό. Ελπίζω να το λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ κύριο Χουντή, παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Καθώ αναμένουμε τι τελικέ προτάσει για τι αερομεταφορέ τη Κομισιόν, ζητάμε ανάμεσα στα άλλα να απαγορευτεί, να σταματήσει κάθε είδου ιδιωτικοποίηση στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Τούτη την περίοδο, στην Ελλάδα, μετά την επιβολή του εκβιαστικού μνημονίου, η κυβέρνηση προχωράει στο ξεπούλημα 14 περιφερειακών αεροδρομίων τεράστιας τουριστικής σημασίας με την έγκριση και την πίεση της Κομισιόν και του Eurogroup αυτό περνάνε στη δικαιοδοσία της Frankfurt που είναι ιδιοκτησία του γερμανικού δημοσίου και της Lufthansa. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε έναν οικονομικό υπεριαλισμό και μια οικονομική ταπείνωση της Ελλάδας αφού με τις συμβάσεις που θα υπογραφούν η Fraport θα έχει το πάνω χέρι στην ελληνική τουριστική αγορά θα δεσμεύσει την ελληνική περιουσία για 40 χρόνια, θα δεσμεύσει το ελληνικό δημόσιο σε απικιακού τύπου συμβάσει και θα έχει τελικά και το πάνω χέρι στην τιμολογιακή πολιτική των υπολείπων κρατικών αεροδρομίων. Ο ελληνικό λαό μαζί με την αυριανή απεργία, γενική απεργία στην Ελλάδα αγωνίζεται να υποχρεώσει την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να υποτάσσεται στα απικιακού χαρακτήρα αιτήματα των δανειστών. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Onorevole Piper, un minuto e 1,5 λεπτό ο κύριος Πίπερ. Θέλω να χαιρετήσω και το κοινό που βλέπω πολύ κόσμο στα θεωρία. Είναι μια συζήτηση ιδιαίτερα εξειδικευμένη με την αρμόδια επίτροπο και ακριβώς οι βουλευτές είναι μέλη των συγκεκριμένων επιτροπών, ιδιαίτερα της Επιτροπής Μεταφορών που ασχολείται με το μέλλον της, α, α, της αεροπορίας της πολιτικής. Σιγά σιγά θα γεμίσει η αίθουσα λόγω των ψηφοφοριών. Για 1,5 λεπτό, κύριος Πίπερ. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στις ε, ευρωπαϊκές ε, αερομεταφορές δεν είναι πάρα πολύ καλή και στον τομέα της απασχόλησης και στον τομέα των εσόδων και στον τομέα του περιβάλλοντος ε, δυστυχώς οι συνέπειες είναι δραματικές. Έχουν χαθεί 20.000 θέσεις απασχόλησης. Και γι' αυτό ο κλάδος των αερομεταφορών στην Ευρώπη έχει ανάγκη από αυτό που θα ονόμαζα μία επανάσταση πλέον. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε τις τάσεις οι οποίες οδηγούν σε αποχωρήσεις εταιριών ουσιαστικά και η κυρία Μπούλτς θα πρέπει να ελέγξει μέσω του δικαίου για τον ανταγωνισμό να μας πει αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα δεν φτάνουν ανακοινώσεις, απαιτούνται νομοθετικές προτάσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν επίσης και τα θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν θα πρέπει εμείς να έχουμε μια νοοτροπία παθητική σε σχέση με όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω εάν πέρα από τις μονομερείς αν θέλετε προβλέψεις θα μπορούσαμε να πάρουμε μέτρα τα οποία να συναντήσουν μια ευρύτερη αποδοχή και να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτά τα οποία η Ευρώπη σε αυτά, να προχωρήσουμε σε αυτά που είμαστε καλοί ε, στις αερομεταφορές. Ευχαριστώ. Βγέλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την Επίτροπο. Πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό, συμφωνούμε. Και νομίζω ότι είμαι μία από τι λίγες λίγε που εκπροσωπούν τον τουριστικό κλάδο στο κοινοβούλιο αυτό. Είναι η δική μου, ο ειδικό μου τομέα αυτό, που εκπροσωπεί δύο εκατομμύρια εταιρείε και εκατομμύρια εργαζομένου. Ο κλάδο του τουρισμού οι αερομεταφορέ, τα ξενοδοχεία, όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι φορείς του κλάδου αυτού ξέρουν ότι η Ευρώπη είναι ο ένα προορισμό στον κόσμο. Αυτό όμω μπορεί να ανατραπεί τα επόμενα χρόνια, γιατί ανακύπτουν διάφοροι φραγμοί. Πρώτα απ' όλα ένα σύστημα που συζητάμε για την διευκόλυνση έκδοση θεωρήσεων και το σχετικό καθεστώ και μετά οι κανόνες για τις τουριστικές θεωρήσεις. Ένας πολύ σημαντικός τομέας που μπορεί να εμποδίσει ε, εκατομμύρια Κινέζους να έρθουν στην Ευρώπη λόγω χάρη. Ευχαριστούμε ο κύριος Βαντάλεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει κατά πρώτο να επιδιώξει να είναι αξιόπιστο. Γνωρίζουμε όλοι ότι πρότεινε την δέσμη μέτρων η, κοινωνική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως πρωτού ακούσουμε την Επίτροπο Μπούλτ. είδαμε πολλά σχέδια κειμένων να φτάνουν στα χέρια των βουλευτών. Ε, ουσιαστικά σπαταλήσαμε πάρα πολύ χαρτί. Οι ίσοι κανόνες του παιχνιδιού, ε, οι ίσοι κανόνες ανταγωνισμού για τους αερομεταφορείς, το τι θα γίνει στην Ευρώπη σε σχέση με τη Μέση Ανατολή με τις αεροπορικέ εταιρείε, η ασφάλεια κατά τις αερομεταφορές είναι στοιχεία που πρέπει να τα δούμε με προσοχή. Και πρέπει επίσης να αποφύγουμε και τις πρακτικές ε, dumping. Θα σας ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση για τις προτάσεις σας στη δέσμη αυτή μέτρων. Ευχαριστούμε κύριο Ρικέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η πρόταση ψηφίσματος που στηρίζουμε δείχνει ότι το Κοινοβούλιο ε, έχει ιδιαίτερο πάθος αλλά και εμπιστοσύνη στο μέλλον αυτού του τομέα, του τομέα των αερομεταφορών. Μας ανησυχούν βεβαίως κάποια στοιχεία όπως τα δικαιώματα των επιβάτων, η τα δικαιώματα του πληρώματος. Εδώ το ε, Συμβούλιο δεν επιτρέπει να προχωρήσει όπως θέλαμε η νομοθεσία περασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα κάποιων κρατών. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το αναχαιτήσουμε. Επίση, έχω την εξή ερώτηση. Τη στιγμή που αναθέτουμε νέε αρμοδιότητε στον Οργανισμό Αεροπορική Ασφάλεια, δεν θα πρέπει η Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποφύγουν τι περικοπέ στον προπολογισμό τη. Στον προπολογισμό του οργανισμού αυτού, επίση, η συμμετοχή μα στην ανάπτυξη των αερομεταφορών είναι ένας πολύ σημαντικό μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη αλλά με τα νέα πιστοποιητικά που ζητούνται ε, δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε χωρίς λόγο τον τομέα, αλλά να τον ενισχύσουμε την κοινοτομία και την έρευνα. Ευχαριστούμε κύριο Δεγκράντε Πασκουάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για την παρουσία της. Και βέβαια πρέπει να πούμε θετικά λόγια για το ψήφισμα, για το περιεχόμενό του. Χρειάζεται όθεση ο τομέα αυτό ε, για να μπορέσει να καταστεί βιώσιμο ε, και ανταγωνιστικό. Η ενίσχυση των αεροπορικών ε, εταιριών, των αερολιμένων και τη αεροναυπηγική βιομηχανία τη Ευρώπη είναι σημαντικό. Τρει ομάδε έχουν με το ψήφισμά του διαγνώσει έγκαιρα τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, όμω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αμοιβαιότητα σε σχέση με τις τρίτες χώρες πρέπει να κάνουμε προβλέψεις για ένα τομέα που ε, προσφέρει ποιοτικέ θέσεις εργασίας. Τέλος, ε, ε, δεν γίνεται να μιλάμε για την ασφάλεια και συνεχώς να χρειάζονται να ενισχυθούν περισσότερα αυτά τα μέτρα. Υπάρχει όμως ένα θέμα που δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Σημείο 28. Για την ισπανική αντιπροσωπεία του ΕΛΚΑ, ε, χωρίς με να κατονομάζεται το Γιβραλτάρ, γνωρίζουμε ότι έχει να κάνει με τη χρήση του ε, ε, του Γιβραλτάρ. Υπάρχει ένα μπλοκάρισμα, είναι απαράδεκτο και το ζήτημα αυτό είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, κυρία Επίτροπε. Επομένως, ε, ούτε το Συμβούλιο ούτε η Κομισιόν έχουν λόγο πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα δύο κυρίαρχων κρατών Ισπανίας και Βρετανίας που συνεχίζουν με το διάλογο, προσπαθούμε να επιλύσουμε τις παλές μας αντιπαραθέσεις και διαφορές. Το θέμα αυτό όμως δεν πρέπει ε, να μπει σε αυτό το ψήφισμα. Και βέβαια ε, θα το λύσουμε με τη Βρετανία που ελπίζουμε να παραμείνει στην Ευρώπη. La parola all'onorevole Ο κύριος De Η κυρία De Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είναι πολύ ε, σημαντικό, πολύ σύντομα να έχουμε μια πλήρη δέσμη μέτρων ε, για, την, ε, για τις αερομεταφορές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του τομέα και να ενισχύσουμε τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια. Υπό το φως της, της προβλεπόμενης αύξησης της κυκλοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων που επιδιώκουμε, πρέπει να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει σύντομα να εγκριθεί η πρόταση κανονισμού για τις θηρίδες στα αεροδρόμια και τις χρονοθυρίδε θα πρέπει να προβλέψουμε την ενίσχυση του ε, ενίου ευρωπαϊκού ουρανού, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή χρήση του εναέριου χώρου και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όλων των φορέων. Η θετική αποτίμηση, ε, ε, μάλλον εξέλιξη του, της δέσμης αυτής μέτρων θα πρέπει να λάβει υπόψη και τους, τις ανάγκες του κλάδου των αερομεταφορών για τον καλύτερο προγραμματισμό των ε, ταξιδιών. Δεν θα πρέπει όμως να υποβαθμιστούν κοινωνικό πρότυπα και η ασφάλεια ε, και αυτά να μην τα ξεχάσουμε γιατί πολύ συχνά έχουμε και σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο. Ευχαριστούμε ο Ζλωτόφσκι για ένα λεπτό. Ε, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όλο και περισσότεροι επιβάτες ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα δείγμα επιτυχίας των αεροπορικών εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο πολλές επιλογές, πιο ελκυστικές τιμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θέλει να αντιμετωπίσει και σωστά μια σειρά από προβλήματα που παραμένουν και θέλει να προβλέψει σε αυτό το πακέτο για τις ενέργειες μεταφορές το μέλλον της αεροπλοεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς αυτό βέβαια να επιβαρύνει υπερβολικά, γραφειοκρατικά, διοικητικά τις αεροπορικές εταιρείες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κυβερνητών, των επιβατών των υπηρεσιών εδάφους πρέπει να απαλληφθούν τίποτε απειλές μπορεί να επιτρέμονται στις αεροπορικές μεταφορές. Χρειάζονται συστήματα αποτελεσματικά για τον έλεγχο των ενέργειων μεταφορών. Καλύτερες επίσης επενδύσεις χρειάζονται για τις υποδομές στα αεροδρόμια και στους τρόπους επικοινωνίας, μεταξύ, στους των συγκοινωνιών μεταξύ αεροδρομίων και πόλεων. Στην ευρωπαϊκή αγορά εναερίων μεταφορών δεν πρέπει να επιτρέψουμε αθέμητο ανταγωνισμό από μεταφορείς που έχουν απαράδεκτες συνθήκες μεταφορών. Σε αυτά όλα πρέπει να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και η Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια νέα ευκαιρία με αυτή τη δέσμη για την αεροπορική βιομηχανία για να δείξει ότι μπορούμε ε, πάνω από τα ειδικά συμφέροντα ορισμένων χωρών, να εκμεταλλευτούμε τι ευκαιρίε ε, που διανοίγονται για του επιχειρηματίε επιχειρήσει και του πολίτε μα. Ε, και γι' αυτό χρειάζεται να υλοποιηθεί οριστικά ο ενίο ουρανός, ε, γιατί αυτό το μέτρο μπορεί να συμβάλλει τα μάλα στη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των αεροπορικών εταιριών τη Ευρώπη, Μόνο έτσι σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά μπορούμε να αποφύγουμε τον εξωτερικό αθέμητο ανταγωνισμό σε αεροπορικέ εταιρείε και κατασκευέ ε, ε, εξαρτημάτων ε, και αεροσκαφών και να αποφύγουμε τις εσωτερικές κακές πρακτικές. Θα πρέπει επίσης, κοιτώντας προς τα εντός, να μειώσουμε το διοικητικό άχθος, να ενσωματώσουμε τις αεροπορικές μεταφορές στις υπόλοιπες μεταφορές με ένα εισιτήριο, να συνδυάσουμε με άλλους τρόπους μεταφοράς τις αεροπορικές, να περιλάβουμε τα περιφερειακά αεροδρόμια στις προσφορές και επίσης να προωθήσουμε σε όλα τα επίπεδα την καινοτομία. Περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον τι προτάσει, κύριε Επίτροπε. La parola all'onorevole Λουκασέφσκα. Λουκασέφσκα, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, ο τομέα των ενέργειων μεταφορών βεβαίω και συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, την διαθέσιμη εργασία, την ανάπτυξη του τουρισμού, των τουριστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη επαφών μεταξύ των πολιτών, τη συνοχή των περιφερειών, την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας των ενέργειων ε, μεταφορών αντιστοιχεί σε 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 360 δισεκατομμύρια ευρώ που συμμετέχουν στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά όλα δείχνουν τη σημασία για το παρόν και το μέλλον του τομέα των ενέργειων μεταφορών. Ωστόσο υπάρχουν αρκετέ δυσκολίε που αντιμετωπίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τομέα αυτό και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε δράση με στόχο. Αφενός μεν την ανάπτυξη θεμητού και δίκαιου ανταγωνισμού, την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών, και αυτό σημαίνει ασφάλεια για ολόκληρο το σύστημα, και βέβαια την προστασία των δικαιωμάτων τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων. Ταυτόχρονα πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου των εθέρων, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τον ευρωπαϊκό μεταφορέα όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Γιατί αυτό επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε ότι θα αναλάβει τα μέτρα που επιβάλλονται στην περίπτωση αυτή. Είμαστε πεπισμένοι ότι τα μέτρα που προβλέπει το ψηφισμά μας θα επιτρέψει μια μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική στρατηγική για όλων των τομέων των αέριων μεταφορών. Ευχαριστώ. Σεχναλόβα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ στο θέμα αυτών των προτάσεων μέτρων. Όλοι ξέρουμε ότι οι νερέ μεταφορέ ε, είναι από τους τομείς τους πιο απελευθερωμένους, απορριθμισμένου στην, ε, στον κόσμο με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τους ε, επιβάτες μεν, αλλά και μειονεκτήματα στις εργασιακές σχέσεις για τους εργαζομένους. Υπάρχουν διάφορες και νοτόμες μορφές απασχόλησης και δεν μπορούμε να υποβαθμίζουμε και να υποτιμούμε τις κοινωνικές πτυχές για τους εργαζομένους. Κυρίως όταν αυτές συνεπάγονται δυσμενείς εξελίξεις για την ασφάλεια των επιβατών. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη για το μέλλον της ενέργειας των ενεργειών μεταφορών. Ο κύριος Ντάλτον έχει το λόγο. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Οι αερομεταφορέ είναι σημαντικέ για την οικονομική ανάπτυξη. Οι Jet και η Ryanair έχουν κάνει πολλά για την περιφερειακή ανάπτυξη από ό,τι έχουν κάνει τα περιφερειακά ταμεία και τα κονδύλια. Αυτό ε, είναι ένα πολύ σημαντικό λοιπόν κλάδο και επίση είναι και παγκόσμιο επίση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να επιτρέπουμε τον δίκαιο Θα πρέπει να επιτρέψουμε για την ε, σωστή λειτουργία των αερομεταφορέων ε, σωστούς κανόνες με τον ε, ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, σαφή προγράμματα και ε, συνολικές συμφωνίες αερομεταφορών με τους εταίρους μας εκτός Ευρώπης. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως το Birmingham που βρίσκεται στην εκλογική μου περιφέρεια. Οι αερομεταφορές δεν είναι απαλλαγμένοι από τους φόρους είναι πολύ ψηλή η φόρη, ε, γύρω στα 170 λίρε για τα Βρετανικά αεροδρόμια, είναι μόνο 42 ευρώ για την Γερμανία. Εδώ έχουμε πολλέ φορέ αθέμητο ανταγωνισμό, γι' αυτό θα πρέπει να επιδιώξουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και όχι αδιάλακτοι. Βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια αγορά και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι ανάγκε μα. Ε, ευχαριστούμε. Ο κύριο Φαν Μίλτεμπουργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημείο που αναφέρεται στο ψήφισμα συγκεκριμένα στα δικαιώματα των επιβατών. Η οδηγία 261. Ε, τη γνωρίζουμε, αλλά υπάρχει σε επίπεδο Συμβουλίου αδιέξοδο. Ξέρουμε ότι υπάρχει το ζήτημα μεταξύ Ισπανίας και Βασιλείου αλλά ε, αυτό το λεπτό ζήτημα δημιουργεί καθυστερήσεις και είναι σε ομοιρία πλέον ε, όλοι. Οι αεροπορικές εταιρείες και οι πολίτες θέλουν ε, όμως σαφήνεια σε ό,τι αφορά και τα δικαιώματά τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα προβεί σε κάποιες ερμηνευτικές, σε κάποια ερμηνεία αυτών των νέων κανόνων. Δεν με βρίσκει σύμφωνη αυτή η προσέγγιση. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ασκηθεί πίεση στο Συμβούλιο ώστε να εγκριθούν επιτέλους οι νέοι κανόνες γιατί μόνο με νέους κανόνες ε, θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου που είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα ιδίως τους συναδέλφους μου ε, και η Προεδρία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δοθεί συνέχεια σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε Μπακ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας, ιδιαίτερα για τη δεσμή μέτρων ε, για τις ενέργειες μεταφορές. Συμφωνώ μαζί ότι χρειάζεται να δοθεί υποστήριξη και κίνητρα έτσι ώστε οι αεροπορικέ εταιρείε, τα αεροδρόμια και το τομέας να ενισχυθεί και να βρεθεί σε πιο ισχυρή θέση. Για όλα αυτά, όπω είπατε και εσεί, χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Πολλέ θέσει εργασία εξαρτώνται άμεσα από τι ενεργέ μεταφορέ εκατομμύρια θέσεις εργασίας που συνεπάγονται την ανάγκη για πολύ σοβαρή αντιμετώπιση της κατάστασης. Συμφωνούν σε αυτό όλοι οι συνάδελφοι. Βεβαίω, δεν πρέπει να λησμονούμε και την κοινωνική διάσταση. Οι συνθήκε εργασία έχουν άμεσε συνέπειε στην ασφάλεια των πτήσεων και πρέπει να αποτελούν άμεση προτεραιότητα στην ε, ασφάλεια των αέριων μεταφορών. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν καταγραφεί έχουν απαριθμηθεί και χρειάζεται να έχουμε υψηλή κατάρτιση και με υψηλά κίνητρα εργατικό δυναμικό στον τομέα των ενέργειων μεταφορών, με κοινωνικό διάλογο, με σαφή ε, ε, ορισμό τη έδρα βάση, της ε, αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τους εργαζόμενους με μεγάλη κινητικότητα. Δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν οι νοοτροπίες των πολύ, των πολύ φθηνών εργατικών αεροπορικών ε, μεταφορικών εταιριών και πρέπει να ενισχύσουμε τις συνθήκες εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Νίλσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περιμένουμε με ανυπομονησία την πρόταση αυτή που θα λάβουμε σύντομα από εσά. Τα τελευταία χρόνια είδαμε πώς ε, ο χώρος ε, εργασίας των τομέα των αερομεταφορών έχει γίνει λίγο σαν την δύση, με συνθήκες εργασίας ε, πολύ κακές, με dumping και, χαμηλού και χαμηλούς μισθούς απαράδεκτα χαμαλού ε, μισθού. Αυτό επηρεάζει και την ασφάλεια από το πρόθεσμα. Χρειάζεται λοιπόν για να αναθετήσουμε αυτέ τι τάσει να υπάρξουν νομοθετικά μέτρα. Και χρειάζεται και ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον κλάδο αυτών. Ε, δεν μπορούμε να ξεχνάμε και να παραγνωρίζουμε τις, εργασίες, τις εργασιακές ε, σχέσεις και ανάγκες των εργαζομένων για εθνικά συμφέροντα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν εδώ αυστηροί κανόνες. Και υπάρχει και ένα θέμα που αφορά και την κοινή γνώμη την οποία βλέπει πολύ θετικά, δηλαδή την ενίσχυση τη ΕΑΣΑ, τη Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν τέτοιε συνθήκε εργασία που να μην επιδεινώνονται ε, συνεχώ και αυτό να αναχαιτήσουμε. Ευχαριστούμε. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε τη δυνατότητα και πάλι να συζητήσουμε μια συνολική δέσμη μέτρων, έτσι ώστε να έχουμε πιο συνεκτική νομοθεσία και όχι με μονομένα μέτρα. Γιατί υπάρχει κίνδυνος με μονομένα μέτρα να είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους και αντιφατικά. Είναι κάτι το οποίο είδαμε και με τον τομέα των συνδρομικών μεταφορών. Ελπίζω στο, μέτρο, στο, μέσο, στο μέλλον λοιπόν η δέσμη μέτρων για τις ενέργειες μεταφορές να οδηγήσει σε μια γενική λύση και αργότερα να ακολουθήσει και ένας τομέας, και μια πρόταση για τον τομέα των αυτιλιακών μεταφορών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν ο τομέα των ενεργών μεταφορών και γι' αυτό πρέπει να μην ε, επιμένουμε σε εθνικά μέτρα ή μεμονωμένα μέτρα, αλλά να βρούμε μια παγκόσμια λύση, μια λύση η οποία θα υποστηριχθεί και από την ΕΚΑΟ, από την Διεθνή Οργάνωση για τις ενέργειε Μεταφορές. Μια παγκόσμια ρύθμιση η οποία μπορεί να δώσει πολύ καλές λύσεις για τις ενέργειε μεταφορές και χαίρομαι που το ψήφισμα μας ιδιαίτερα ε, δίνει έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε να είναι πιο ανταγωνιστικές οι εταιρείε μας σε σχέση ιδιαίτερα με τις ανταγωνιστικές πιέσεις από τις χώρες του Περσικού κόλπου και τις αντίστοιχε εταιρείε. Χρειάζεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει τα ζητήματα αυτά και να καταθέσει τις προτάσεις της και τις ε, προτάσεις τροποποίησης στο πλαίσιο αυτής της θέση μέτρων. Ιδιαίτερα δε καλό και τα κράτη-μέλη, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει ρυθμίσεις μόνο αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο των εναέριων μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Σιμών. Σάιμον. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το πρόβλημα των μεταφορών για χρόνια είναι ότι συνεχίζουμε να τα αντιμετωπίζουμε σε ένα τομέα και θέτουμε ερωτήσει γι' αυτόν, αντί να σκεφτόμαστε πώ θα ταιριάξει με τι ανάγκε τη οικονομία και τη κοινωνία συνολικά. Γι' αυτό έχουμε προκύψει, έχουν προκύψει τέτοιε γελίε καταστάσει όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει χτιστεί ένα 77ο αεροδρόμιο στο Λονδίνο, ε, γελίε αποφάσεις, ενώ πρέπει να στηρίξουμε περιφερειακά αεροδρόμια όπω το Μπέρμιχαν, το οποίο φέρνει ένα δις ε, στερλίνε εισόδημα στην τοπική οικονομία. Φανταστείτε πόσο συμβάλλει στην εθνική οικονομία, στον εθνικό κορβανά και κατά πόσον θα έπρεπε να ενισχυθεί. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε την στρατηγική των αεροδρομίων μας ε, συνολικά, σφαιρικά και επίσης και τις εργασιακές συνθήκες των ε, ανθρώπων αυτών. Ε, οι μηδενικές συμβάσεις, ε, το σύστημα pay to fly δεν μπορούν να συνεχιστούν αδιάκοπα. Πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Μοντέρο κυρία Μοντέρο Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, ε, συνάδελφοι. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις που περνάει ο κλάδος των στην Ευρώπη. Εδώ και χρόνια οι αεροπορικές εταιρείες, η ε, αεροναυπηγή και την οποία συζητάμε, είναι στοιχεία του κλάδου αυτού, όπως και τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια όμως Πολλές φορές αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό αδάσταχτο και πολλές φορές αθέμητο από τρίτες χώρες. Εδώ και χρόνια, ε, λόγω των κανόνων τη Ευρώπη τα αεροδρόμια δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, την ε, διόγκωση κυκλοφορία σε μη ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και τι αλλαγέ στι διαδρομέ κάποιων πτήσεων που έχουν επηρεάσει όλο ιδιαίτερω ε, περιφερειακά αεροδρόμια. Πρέπει λοιπόν αυτή την ευκαιρία να την εγκαταλευτούμε, κυρία Επίτροπε, για να παρέμβουμε και να ε, αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μα. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική για τα περιφερειακά αεροδρόμια εδώ, λαμβάνοντα υπόψη και την ανάγκη τη ενίσχυση από το κράτο για τα αεροδρόμια αυτά και το πώ τα περιφερειακά αεροδρόμια μπορεί να συμβάλλουν και να στηρίζουν ω ραχοκοκαλιά τα κεντρικά αεροδρόμια. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ξεκάθαρη θεώρηση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι τα περιφερειακά αεροδρόμια επιτρέπουν να συνδέονται ε, πρόσωπα, ε, τόποι, ε, αγαθά και υπηρεσίε. Εδώ οι υποδομέ πολλέ φορέ ε, χρειάζονται ενίσχυση, αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτέ είναι πολλέ φορέ και πύλε από τι οποίε περνούν οι τουρίστε. Άρα αυτό στηρίζει τι ε, οικονομίε, τι τοπικέ οικονομίε των περιφερειών τη Ευρώπη. Είναι σημαντικά λοιπόν όλα αυτά για την ε, κοινωνική διάσταση τη Ευρώπη και για εξόχω απόκεντρε περιοχέ όπω η Μαδέρα. Ευχαριστούμε ο κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλέ προκλήσει, κινδύνου και αλλαγέ. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ελπίζουμε να, να μας υποβάλει μια δεσμή φιλόδοξη, λαμβάνοντα υπόψη τι ανάγκε βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορούμε πλέον να παραμελούμε το πώ επιτρά ε, ε, η κυκλοφορία των μεταφορών στο κλίμα, όπω επίση δεν γίνεται με την εκπομπή ε, διοξιδίου του άνθρακα και αερίων του θερμοκηπίου. Η πολιτική αεροπορία πολλέ φορέ αναγκάζεται να λειτουργήσει με αυξημένε ανάγκε, ενώ έχουμε αυστηρού στόχου για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ε, μέσα στο 2016. Το ίδιο περιμένουμε να γίνει και με την διάσκεψη των ημερών στο Παρίσι, την COP21. Πώ θα πετύχουμε λοιπόν μια τέτοια μείωση, οι τεχνολογικέ εξελίξει, οι ε, αεροπορικές στάσεις ή τα ολοκληρωμένα εισιτήρια είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ξαναδούμε, να δούμε τις ανάγκες του τομέα για να στηρίξουμε την ε, δομή των ευρωπαϊκών αερομεταφορών και να επιτρέψουμε στα κάτι μέλη να βελτιώσουν τις υποδομές των ευρωπαϊκών αεροδρομίων, ώστε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο με ευνοϊκού όρους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Βλασίκο Βαμπένοβα. Κυρία Επίτροπε, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ο τομέα. Αντιστοιχεί σε πάρα πολλές θέσει εργασία. 10 εκατομμύρια πτήσεις κάθε χρόνο στην Ευρώπη, 500.000 εργαζόμενοι στην, στον κλάδο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει. Και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η σταθεροποίηση των εναέριων μεταφορών και για την απελευθέρωση βεβαίω έχει πολύ μεγάλη σημασία εξασφάλιση υψηλού επίπεδου υπηρεσιών και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών. Αυτό άλλωστε αποτελεί και παράγοντα που λαμβάνει υπόψη του για την επιλογή μιας πτήσης του επιβάτης. Επίσης, πολύ σημαντικό μέλημα είναι η ασφάλεια των μεταφορών αυτών. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε να ε, επιβαρύνονται με δυσμένες συνθήκες οι επιβάτες, γιατί σε ορισμένα αεροδρόμια βλέπουμε πολύ δυσμένες συνθήκες. Ευχαριστούμε, Γιονγκέριους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και Επίτροπε. Τον προηγούμενο Μάη το Πανεπιστήμιο της γάντης έκανε μία μελέτη που ε, καταδεικνύει ότι τα μισά αεροπλάνα της εταιρεία του Μπακού. Τα κυβερνούν πολύ νέοι κυβερνήτες με συμβάσεις pay to fly. Έχουμε και με σημαίες ευκαιρίας, ε, έχουμε ε, κάποιες άλλες ε, συμβάσεις και όλα αυτά συνεπάγονται δι, μεγάλο κίνδυνο και ρίσκο. Είναι επισφάλιση συνδικές εργασίας. Και είναι και αθέμητες και ε, επονδύσεις αυτές οι πρακτικές των επιχειρήσεων. Τι θα κάνετε να καταπολεμήσετε αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό, κυρία Επίτροπε. Σίγουρα το πρόβλημα δεν λύνεται από μόνο του, αλλά εσείς, Επίτροπε, τι μπορείτε να κάνετε ε, και για να προωθήσετε τις διεθνείς μεταφορές τι θα γίνεται με τα δικαιώματα προσγείωση, θα πρέπει να εξαρτώνται από καλέ συνθήκε εργασία των εργαζομένων. Ευχαριστώ κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Η μελλοντική δέσμη για τι ενέργειε μεταφορέ αποτελεί μια έκλεκτη ευκαιρία για βελτίωση των συνθήκων τη ΕΑΖΑ, τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Ενέργειων Μεταφορών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαφυλαχθεί και ο τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ο κλάδος της κατασκευής. Έχουμε 4.000 εργαζόμενους ε, σε άμεση σχέση εργασίας και χιλιάδες άλλους στην αλυσίδα προμηθειών, στη δική μου μόνο εκλογική ε, περιφέρεια. Αλλά υπάρχει ακόμη μεγάλη καθυστέρηση ως προς την πιστοποίηση αεροσκαφών λόγω των δυσκολιών που έχει η ΑΖΑ στη διαχείριση των φακέλων αυτών. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να επανεξεταστούν Πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε ένα παγκόσμιο σκηνικό και πάνω απ' όλα το λέω και ως μέλος της Επιτροπής των Προϋπολογισμών, δεν πρέπει να επιβαρυνθεί περισσότερο με ε, δαπάνες ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν σας καλώ να βοηθήσετε να ε, λειτουργήσει αποτελεσματικά υπέρ του κλάδου η ΕΑΣΑ και να βελτιώσει ιδιαίτερα με τις πολύ καλές επιδόσεις που έχει ήδη την ασφάλεια των πτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να περάσουμε στη διαδικασία Catch Πρώτα απ' όλα, η κυρία Κλούινα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τον Πρόεδρο και την Επιτρόπο Μπούλτς και προσβλέπω να ε, ενημερωθώ τον επόμενο μήνα για αυτή τη δέσμη μέτρων για την αεροπορία που ε, με την απελευθέρωση έχει ε, προσφέρει ωφέλη και πλανεκτήματα και στις εταιρείε και στους πολίτες. Βέβαια σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε και αρνητικά στοιχεία και θετικά οι συγχωνεύσεις, οι νέες εταιρείε περιφερειακές έχουμε τη Ryanair, την EasyJet. Ε, το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν και προβλήματα. Δεν προχωρά ο ενιαίος ε, ουρανός, ε, τα σλότ, οι χροθυρίδες και τα δικαιώματα των επιβατών. Εκεί έχουμε προβλήματα. Πρέπει σίγουρα να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών. Ένα άλλο που θέλω να χαιρετήσω είναι ε, η συνεργασία μας ε, με εταιρείες από άλλες ε, χώρες, χώρες της Βαλτικής για παράδειγμα, σίγουρα είναι καλό να έχουμε με άλλες αεροπορικές εταιρείες συμφωνίες, γιατί ήρθαν να παραμείνουν αυτές οι εταιρείες, τις χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι επιβάτες και θα πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία ενός οχυρού τείχους γύρω από την Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε επομένως συμφωνίες με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Δεν μπορούμε να φαλοσκοπούμε. Είναι παγκοσμιοποιημένο ο τομέα αυτό και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και προ όφελο των καταναλωτών μα και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαρία. Κύριο Μαριά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αεροναυπηγική βιομηχανία είναι ένα από του σημαντικότερου συντελεστέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη και την απασχόληση ενώ παράλληλα συνδέεται στενά με τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών στην ευρώπη με κύκλο εργασιών εκατό δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και μισό εκατομμύριο περίπου άμεσες θέσεις εργασίας. στην ελλάδα η τρόικα και η μνημονιακή συγκυβέρνηση παραχώρησαν κατ' εντολή της μέρκελ για 40 συν 10 χρόνια 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην κρατική γερμανική εταιρεία Fraport, η οποία εκμεταλλεύεται επίσης και τον αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος μια κρατική εταιρεία λοιπόν αποκτά κυρίαρχη θέση στην εκμετάλλευση αεροδρομίων στην ευρώπη και κατακτά επίσης κυρίαρχη μονοπωλιακή θέση στην ελληνική τουριστική αγορά κατά παραβίαση των κανόνων της ευρωπαϊκής ένωσης περί ελεύθερου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων. έτσι τα ελληνικά αεροδρόμια γερμανοκρατούνται και ο ελληνικός τουρισμός μετατρέπεται πλέον σε γερμανικό τσιφλίκι και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. ευχαριστώ. Ο κύριος Φροντζούλικα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, συνάδελφοι. Συμφωνώ με όλες τις προτάσεις ε, της δεσμής μέτρων ε, για το μέλλον των ευρωπαϊκών αερομεταφορών γιατί θα στηρίξει τον κλάδο αυτό, την ανταγωνιστικότητά του, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τα αεροδρόμια και την ε, εταιρεία, την, ε, τον κλάδο των αεροναυπηγικής. Ε, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στην, ε, στην διεθνή παγκόσμια αγορά και να έχουμε και στόχους βιωσιμότητας. Θα πρέπει να έχουμε καινοτομία και στον ε, χώρο της ενέργειας, του ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας, των, της ψηφιοποίησης και να αναζητούμε σύγχρονες λύσεις. Γι' αυτό ε, πρέπει να υπάρχουν και περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως μέτρα που να φασίζονται στις ανάγκες της αγοράς, για να αντιμετωπίσουμε ε, το θέμα των εκπομπών ε, αερίου του θερμοκηπίου και τους φόρους για τον άνθρακα και να δούμε τις ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία επιτρέπ εφαρμόζοντας την ε, οδηγία για τα τέλη των αεροδρομίων πολύ σύντομα. Ε, επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και για τα περιφερειακά αεροδρόμια εντό τη Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. ΠΑΕΤ. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Η δική μας εταιρεία Estonian Air έχει λάβει κρατικές ενισχύσεις από την ε, κυβέρνηση και πρέπει να τα καταβάλει αυτά από φάση κομισιών και πτώχευσε τελικά η εταιρεία μας. Χάσαμε την ανταγωνιστικότητα, 164 άτομα χάσαν τη δουλειά τους αυτή η κρατική ενίσχυση ε, θεωρείται επιβλαβής για τον ανταγωνισμό. Με γιατί ε, ανταγωνισμό μιλάμε, η Ιστονία έχει πολύ λίγε συνδέσει αεροπορικέ. και πολλέ αεροπορικέ εταιρείες δεν θέλουν καν να πετάξουν από εκεί προ την Ιστονία. Η πτώχευση του εθνικού αερομεταφορέα περιορίζει την ανταγωνιστικότητα και δυσχεραίνει την σύνδεση της χώρας μας με άλλες περιοχές του κόσμου. Πώς λοιπόν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ένωσης αυτή η πολιτική με τη νέα δέσμη μέτρων για την αεροπορία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί ε, με τον ίδιο τρόπο ε, στα περιφερειακά αεροδρόμια. Θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, ώστε και οι μικρές περιφερειακές χώρες να μπορούν να έχουν άμεσες απευθείας συνδέσεις με μεγαλύτερες πόλεις ε, σε άλλε χώρε, γιατί η αγορά από μόνη τη δεν θα τα ρυθμίσει αυτά. La parola all'onorevole Σακοράφα. Κύριε Σακοράφα. Κύριε Επίτροπε, τι νόημα έχει να μιλάμε σήμερα για ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αερομεταφορών, διεθνή συνεργασία, προστέ τιμέ για του καταναλωτέ, κοινωνική ατζέντα και υψηλό επίπεδο ασφάλεια, όταν όλα αυτά δεν λειτουργούν προ όφελο των πολιτών με τι ευλογίε φυσικά του ευρωπαϊκού διευθυντηρίου ή μήπως είναι ένα μονοπόλιο τελικά καλό μόνο όταν είναι κρατικό και γερμανικό. Τι θέλω να πω. Ενώ συζητάμε για το μέλλον των ευρωπαϊκών αερομεταφορών, στην Ελλάδα, όπως υπόθηκε και προηγουμένω, από συναδέλφους, παραχωρούνται 14 κρατικά περιφερειακά αεροδρόμια στη γερμανική κοινοπραξία Fraport Schlendel με ληστρικούς όρους και με την ευλογία και την πίεση της Τρόικα. Μια επιλεκτική αρπαγή μόνο των αεροδρομίων που κρίθηκαν οικονομικά βιώσιμα για τα οποία αόριστα ευαγγελίζεται την αναβάθμισή τους. Στην πραγματικότητα δεν εξασφαλίζει καμία αναπτυξιακή προοπτική αφού δεν αναλαμβάνει καμία σοβαρή επενδυτική δέσμευση μια παραχώρηση θυσία στην εκβιαστική μνημονιακή πολιτική που δημιουργεί ένα απαράδεκτο μονοπόλιο προ όφελο τη γερμανική κυβέρνηση και επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο με αποζημιώσει προ υφιστάμενου προμηθευτέ. Μια παραχώρηση που όχι μόνο δεν κατοχυρώνει του εργαζόμενου, αλλά του θέτει σε καθεστώ εργασιακή ομοιρία. Έτσι εννοεί, κυρία Επίτροπε, την ανάπτυξη Ευρώπη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά μου να μπορώ να μιλήσω και στην μετρική μου γλώσσα, έστω ε, για λίγες φράσεις, αλλά κυρία Επίτροπε, προφανώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι ανάγκε των αερομεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι χρειαζόμαστε ίσω κανόνε ανταγωνισμού. Έπειτα υπάρχει και το αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο αναφέρθηκε εδώ. Ανησυχεί το θέμα αυτό, όπως και το πώς θα έχουμε αρκετά ισχυρά νομοθετικά εργαλεία για να περιορίσουμε τη, τα αέρια του, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Και η εκπρόσωπη του Ευρωκοινοβουλίου στην ε, διάσκεψη του Παρισιού θα πρέπει να προωθήσουν μαζί με τις δικές σας προτάσεις την ε, ανάγκη αυτή ακριβώς οι αερομεταφορές να καλύπτονται από διεθνείς συμφωνίες. Βλέπουμε λοιπόν ήδη να ε, υπάρχει ε, τάση ενίσχυσης των περιφερειακών αεροδρομίων. Ήδη στην Ιρλανδία υπολογίζουμε να αυξηθεί πολύ η κίνηση επιβατών με ένα εκατομμύριο παραπάνω αφήξεις, κάτι που θα στηρίξει οπωσδήποτε την τοπική οικονομία. Γι' αυτό θέλουμε να εφαρμοστεί οδηγία ε, για τα αεροδρόμια. Ευχαριστούμε και τώρα λόγω στην Επίτροπο την κυρία Μπούλτ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι προβουλευτές, ήταν μια καταπληκτική συζήτηση, η οποία καταδεικνύει και σε μένα πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Παρά τις μεγάλες προκλήσεις, γνωρίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε ε, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς. Εν συντομία, να σχολιάσω ορισμένα από ε, τα ερωτήματα και σχόλιά σας. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα, διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, εκτός αν μιλήσω πολύ γρήγορα, αλλά τότε θα δυσκολέψω το έργο των διερμηνέων. Θα προσπαθήσω λοιπόν να καλύψω όσα περισσότερα ζητήματα μπορώ και σας παρακαλώ να μου στείλετε τα πρόσθετα ερωτήματά σας γραπτός, εάν δεν έχω λάβει τις απαντήσεις που θα θέλατε. Πρώτα απ' όλα, το πιο συχνό ζήτημα ήταν ε, η εξασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού. Εμείς ε, συμφωνούμε με το στόχο της εξασφάλισης ε, του θεμητού ανταγωνισμού στον τομέα της αεροπορίας. Και γι' αυτό το σκοπό έχουμε διάφορα εργαλεία. Πρώτα απ' όλα, υγιείς πρακτικές επιλογής, εφαρμογής των μερών συμφωνιών, Επίσης, οι υπηρεσικές συμφωνίες, ιδίως με εμπορικού φορείς, πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να ε, να θεωρήσουμε και τη ρήτρα περί δίκαιου ανταγωνισμού για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη διάταξη αυτή τη διαπραγματεύσεις μας με τρίτες χώρες. Αποκλειστική αρμοδιότητα βέβαια ε, της Κομισιόν και των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού ισχύει και πρέπει να γίνεται σεβαστή σε κάθε περίπτωση. Και αυτό θα το αναφέρουμε ξεκάθαρα. Το επόμενο ερώτημα ήταν οι επιδοτήσεις. Να υπογραμμίσω ότι οι επιδοτήσεις είναι κάτι που προ το παρόν αποτελεί ισχυρισμό. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη και αν υπάρχουν επιδοτήσει ενισχύσει κρατή. Θα πρέπει να δούμε αν ε, βλάπτουν τι αεροπορικέ εταιρείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ε, μα ενδιαφέρει. Να μην λησμονούμε ότι η απώλεια ανταγωνιστικότητα ε, τη αεροναυπηγική βιομηχανία τη Ένωση οφείλεται σε διάφορου λόγου. Παραδείγματο χάρη, κατακαιρματισμό ε, των συστημάτων αεροπορικών μεταφορών και ανελειπής εφαρμογή ε, του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, υπάρχει ε, υποδομέ. και ε, επίπεδο ανταγωνισμού που δεν είναι ισότιμο. Εμείς προσπαθούμε τη στρατηγική μας για την Ευρωπαϊκή να καταπολεμήσουμε αυτά τα προβλήματα. Επόμενα θέματα. Ο κανονισμός. Μέχρι στιγμής Μέχρι στιγμής Ακούστηκαν βέβαια ε, κάποιες, ε, κάποιες, ε, κάποια παράπονα για τις αθέμιτες πρακτικές, αλλά δεν έχουμε διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Εμείς πάντως θα αναθεωρήσουμε τον κανονισμό αυτό. Και ίσως έχουμε μια άλλη πρόταση στις αρχές του 2016 μετά από αυτήν την αξιολόγηση. Σε ό,τι αφορά συνθήκες εργασίας. On a competitive σε μια ανταγωνιστική αγορά η πίεση για τη μείωση του επιχειρησιακού κόστου είναι μεγάλη και αυτό μπορεί να επηρεάσει τα κοινωνικά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Αττικής για την αεροπορία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. Οι διάφοροι φορεί ε, σε όλη την αλυσίδα θα πρέπει να μπορούν να αποφελούνται από το μεγάλο αυτό δυναμικό για να ε, παραμείνει σε ισχύ ε, το θεματόλογο και το κοινωνικό και να δημιουργηθούν ποιοτικέ θέσει εργασία. Σε αυτά τα πλαίσια το σημαντικότερο είναι ένας ισχυρός κοινωνικός διάλογος. Και πιστεύω ότι ήδη έχουμε με τη διάσκεψη των κοινωνικών ζητημάτων στις μεταφορές ε, τον Ιούνιο 2015 θέσει τα θεμέλια για αυτό το διάλογο. πράγματι για το επόμενο θέμα θα πρέπει να έχουμε τις νομικές, ε, τα νομικά στοιχεία για τις εξελίξεις ε, για να δούμε τι γίνεται με τα ατυπικά φόρουμα και τι επιπτώσεις έχει αυτή η πρακτική. Θα έχουμε σύντομα μια μελέτη ε, για τις συνθήκες εργασίας στα αεροδρόμια και επίσης για την ΕΑΣΑ πρέπει να πω ότι έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας για να αξιολογήσει τις πτυχές ασφαλείας των νέων μοντέλων. Κατάρτιση δεξιότητες. Η ασφάλεια στην Ευρώπη ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα και έτσι πρέπει να παραμείνει. Θα πρέπει να δοθεί κατάρτιση, εκπαίδευση, να αποτελεί σε αυτό προτεραιότητα. Έχουμε την Εικονική Ακαδημία της ΆΣΑ, η οποία ε, αναδεικνύεται σε ένα πραγματικό δίκτυο διαπιστευμένων εκπαιδευτικών ε, ιδρυμάτων στον τομέα της αεροπορίας. Τα κοινά πρότυπα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τις ε, σχετικές αρμοδιότητες των επιθεωρητών ασφάλειας, είναι ζητήματα τα οποία επίσης εξετάζουμε. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, έχουμε ισχυρά ρυθμιστικά εργαλεία όπως το ζήτημα για την καταπολέμηση των θερμοκηπιακών αερίων. Σίγουρα ε, θα πρέπει ε, παγκοσμίως ε, να εφαρμοστούν οι στόχοι από το 2020 και για τα αεροσκάφη να υιοθετηθούν οι πρώτοι κανόνες για, τα, για τις εκπομπές αερίων πρόκληση, το πρόβλημα του Γεβραλτάρ αναφέρθηκε εν μέρη. Θέλω να σχολιάσω ε, συντομία, διότι πραγματικά ε, το Γεβραλτάρ κινδυνεύει να ε, υπονομεύσει εργασία ετών και από τα τρία θεσμικά όργανα. Εμείς ε, να αναβαθμίσουμε τη δέσμευσή μας και γι' αυτό ε, καλούμε και τις δύο πλευρές να ακολουθήσουν μια επικοδομητική προσέγγιση για να βρεθεί μια ρεαλιστική λύση. Η στρατηγική για την αεροπορία θα πρέπει να δώσει την πολιτική όθηση για την επίτευξη πρόοδου στον τομέα αυτό. Ιδίω για τα δικαιώματα των επιβατών ε, και το ΑΣΕΣ του 2 που αναφέρατε ορισμένα από εσάς. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει ε, στις αρχές Δεκεμβρίου ε, τη στρατηγική για την αεροπορία. Δεν θα είναι όμως άπαξ το εγχείρημα αυτό, γιατί δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Όμως θα πρόκειται για την απαρχή μιας διαδικασίας η οποία θα μας οδηγήσει, πιστεύω, σε μια ισχυρή ανταγωνιστική αεροπορία και ακόμα πιο ισχυρή η αγορά στον τομέα της αεροπορίας. Προσβλέπω ε, στην συνέχιση της στενής συνεργασίας με όλες και όλους σας και πραγματικά είμαι αισιόδοξη ότι θα το καταφέρουμε και θα έχουμε σύντομα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε να είμαστε ηγέτες ε, στην παγκόσμια αγορά της αεροπορίας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Έχω λάβει επτά προτάσεις ψηφίσματος για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Κλείνει η συζήτηση εδώ και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο και υπενθύμιζω σε όλους τους συναδέλφους. ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί η ένατη εκδήλωση του βραβείου Λουξ, κινηματογραφικού βραβείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που προβάλλει τα καλύτερα φιλμ ανεξάρτητων σκηνοθετών και την κινηματογραφική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι ταινίες που έχουμε φέτος είναι το Mediterranean, το Euroc και το Mustang υποτιτλισμένοι, σε όλες τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν το βραβείο και σας καλώ όλους να παρακολουθήσετε τις τρεις ταινίε και να ψηφίσετε μέχρι τις 23 Νοεμβρίου. Διότι στις 24 έχουμε την εκδήλωση απονομής και θα ήθελα να ενημερώσω έτσι και το κοινό μας, το οποίο βρίσκεται στα θεωρία και παρακολουθεί τη συνεδρίαση, ότι προβλέπεται και ψηφοφορία με συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι θα κρίνουν τις τρεις αυτές ταινίε. Έτσι λοιπόν θα δοθεί και η αναγνώριση από τους κριτές παύλα πολίτες. Πρέπει να πάτε στο Lux Price, στον ιστότοπο και να πατήσετε το σημείο που λέει ψηφίζουμε για την ταινία. Αυτό επιτρέπει νομίζω και τη συμμετοχή των πολιτών στην προαγωγή της κινηματογραφικής παραγωγής της Ευρώπης. Υπενθυμίζω λοιπόν, μέχρι τις 23 οι βουλευτές πρέπει να έχουν ψηφίσει και ελπίζω ως το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές να συμμετάσχουν διότι άλλωστε το ακούσατε όλοι στην αρχή της ε, περίοδου συνόδου η Αντιπρόεδρος Κώστα έκανε την αναγγελία και ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας ώστε δυνατόν λοιπόν περισσότεροι από καλούνται να συμμετάσχουν και να επιλέξουν από τις ταινίες Μεδiterranea, Ούροκ, Μάσταγκ. Τώρα διακόπτω τη συνεδρίαση για να ξαναρχίσουμε στις 7 το βράδυ, ακριβώς με τις ψηφοφορίες.